και να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για τέσσερα λεπτά. Yes, thank you, Chair. Uh, I'm, I'm glad we... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα της διαφανείας και αρχίζω λέγοντας, διαβάζοντας μάλλον κάτι από μια τηλεοπτική σειρά που μου αρέσει το Yes Prime Minister ο Sir Humphrey Appleby λέει στον Πρωθυπουργό ανοιχτή διακυβέρνηση, ελευθερία της ε, Έτσι πρέπει να λέμε πάντα στον τύπο, οτιδήποτε μπορούν να το βρουν και μόνοι τους. Αυτό είναι περίπου, αυτή είναι περίπου και η στάση των ενωσιακών θεσμικών οργάνων σήμερα. Όλοι γνωρίζουμε συνάδελφοι ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών είναι, βρίσκεται σε ναδύρα και πρέπει τώρα να δείξουμε ότι η ευρωπαϊκή θεσμοί είναι πιο διαφανής και έτσι να δώσουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους πολίτες. Γιατί για 50 χρόνια η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση βασίζονταν σε διπλωμάτες και δημόσιους υπάλληλους που δούλευαν μεν εξαιρετικά αλλά αυτό είναι το παρελθόν με δούλευαν με απόρριτα, απόρριτες διαδικασίες. Σήμερα είμαστε σε μια πολιτική ένωση, σε μια Ευρώπη των πολιτών και άρα η διαφάνεια είναι ουσιώδες θέμα της λειτουργίας μας. Λοιπόν, πριν επισέλθουμε σε λεπτομέρειες της έκθεσης που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή ΕΛΕΦ και θα ψηφιστεί αύριο, να σας πω μερικά λόγια για το εναλλακτικό ψήφισμα του ΕΛΚ που με εκπλήσει διότι φαίνεται ο, να μην ζητάει περισσότερη διαφάνεια αλλά τη μειώνει και το βρίσκω εκπληκτικό διότι υπάρχουν και μέλη του ΕΛΚ που προέρχονται από χώρες με παράδοση διαφανείας είναι μάλιστα από τις εθνικότητες που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαφάνεια στην Ένωση. Νομίζω ότι στο σκεπτικό γάμα του ΕΛΚ, του ψηφίσματος του ΕΛΚ, δεν ε, δείχνουν να σέβονται και πολύ την ευφυΐα των πολιτών, διότι λένε ότι είναι τόσο πολύπλοκη η διαδικασία της νομοθετικής έγκρισης ώστε χρησιμοποιούνται μυστικά έγγραφα που είναι τόσο ουσιώδη κτλ είναι σαν να λένε μη στεναχωριέστε το μυαλουδάκι σας δεν είναι για αυτά τα πράγματα και διαβάζω ε, αναφέρω ακόμη μια φορά τη σειρά Yes Prime Minister όπου λέει ο Σερ στον Τζον Appleby μα οι πολίτες μιας δημοκρατίας έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν και απαντάει ο Σερ Χάμφρι όχι έχουν το δικαίωμα να αγνοούν η γνώση σημαίνει συνενοχή ενώ η άγνοια έχει κάποια αξιοπρέπεια. Αυτό βέβαια μπορεί να ε, είναι θεμητό να λέγεται στην τηλεόραση αλλά όχι εδώ σε από πολιτικούς της Ένωσης. Πρώτον λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να αναθεωρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία 1049. Είναι βασικό, είναι απαράδεκτο η Κομισιόν και το Συμβούλιο να μπλοκάρουν τα πράγματα. Δεύτερον η διαφάνεια πρέπει να είναι ο κανόνας και το απόρριτος χαρακτήρας, η μυστικότητα, η εξαίρεση, ενώ τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Έχουμε κάνει μερικές πολύ πρακτικές και ρεαλιστικές προτάσεις, παραδείγματος χάρη κάθε όργανο της Ένωσης και το Κοινοβούλιο, να ορίσει έναν υπεύθυνο διαφανείας. Σήμερα έχουμε τόσο πολλούς δημοσίους υπαλλήλους να βάλουμε κάποιον να ασχολείται με αυτό το θέμα για να δημιουργηθεί επιτέλους μια κουλτούρα διαφανείας. Έπειτα, επειδή έχουμε μεγάλη εμπειρία για τις διαφορές και την επίλυση διαφορών στα δικαστήρια, χρειάζονται κάποιες ελαφρύτερες διαδικασίες για την επίλυση διαφορών ως προς την πρόσβαση στα έγγραφα. Είναι παράλογο να επιβαρύνουμε τα δικαστήρια χρόνια και χρόνια με τέτοιες διενέξεις. Ναι, πρόεδρε, τελειώνω, τελειώνω, τελειώνω. Και τέλος, πρέπει να έχουμε καλύτερες διαδικασίες για τη δαξινόμηση το, του χαρακτήρα των γράφων και τις διαδικασίες των ε, ε, συνεδριάσεων που γίνεται και κλεισμένων των θυρών. Ενώ αυτό σήμερα τα αποφασίζουν οι ψηλόβεθμοι υπάλληλοι. Πρέπει να υπάρξουν άλλα κριτήρια, πιο ανοιχτά και ένα ανεξάρτητο σώμα που να τα παρακολουθεί. Ευχαριστούμε κυρία Σοφία μου και τώρα θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Κοράτσα Μπίλντ. Η δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα είναι καθοριστική, είναι σημαντική για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ αυτών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολίτε έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται για αυτούς, για τους πολίτες και να υπάρχει λογοδοσία, ούτως ώστε τα δημόσια χρήματα να ξοδεύονται σωστά. Είναι σημαντικό να υπάρξει πλήρης δέσμευση στην αρχή της διαφάνειας και το κοινοβούλιο, θα πρέπει, το κοινοβούλιο βρίσκεται πραγματικά στην πρώτη γραμμή. Οι περισσότερες ε, ε, συζητήσεις εδώ δημοσιοποιούνται. Ε, Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα. Γι' αυτό που απευθύνει μια έκκληση προ χώρε μέλη, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προχωρήσουν με τον κανονισμό, ούτως ώστε να βελτιωθεί η δημόσια πρόσβαση στα κείμενα όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Α ανοίξουμε τι πόρτε μα, α ενισχύσουμε του πολίτε να συμμετάσχουν περισσότερο για να αποκτήσουν την αίσθηση ότι είναι τμήμα μια ευρύτερη κοινότητα, όπου οι αποφάσει λαμβάνονται για του πολίτε με έναν δημοκρατικό τρόπο συνεργαστούμε για μια πιο δημοκρατική και διαφανή Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, κυρία Μαρία Κοράτσα Μπίλτ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Κάστρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να συγχαρώ τη Σόφη για την εξαιρετική της δουλειά και πραγματικά χαίρομαι που συνεχίζει την αναθεώρηση που προσπάθησα και εγώ να φέρω πέρα εκ μέρους του Κοινοβουλίου. Παρά τις συμβαστικές λύσεις που βρήκε το Κοινοβούλιο βεβαίως, το θέμα αυτό έχει μπλοκαριστεί και στο επίπεδο του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζω όμως ότι με την έκθεση αυτή θα πάμε ένα βήμα παραπέρα. Και επιτρέψτε μου Σόφη, είναι αρκετά avant-garde, είναι πολύ προχωρημένη η έκθεση αυτή γιατί στέλνει ένα μήνυμα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο που λέει ότι το Κοινοβούλιο αντί να οπισθοχωρεί δεν ακολουθεί τροπαθέστερη ε, στάση αλλά απαιτεί να υπάρξει διαφάνεια και άνοιγμα της πρόσβασης όλων στα έγγραφα. Είναι πραγματικά ντροπή που το ε, ΕΛΚ προσπαθεί να υπονομεύσει το έυρος της ε, έκθεσης αυτής και το στόχο της. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι περισσότερη διαφάνεια, όχι λιγότερη. Και το λέω επανειλημμένος, το είπα στην κυρία Σόμερ. Τι φοβάστε γιατί φοβάστε να ε, ενημερώσετε τους πολίτες σας εφόσον αυτούς εκπροσωπείτε. Εάν φοβάστε τη δημοκρατία παρατήστε αυτή τη δουλειά και βρείτε κάποια άλλη. Διότι η λογοδοσία είναι η ουσία της δημοκρατίας πρέπει εδώ να δούμε ένα από τα βασικά προβλήματα τα οποία δεν τα έχουμε συζητήσει ακόμα. Αυτό είναι το βάρος που ασκείται στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις με τις διαρκείς και συνεχείς απαιτήσει που υπονομεύουν και τη δική τους δουλειά και την ικανότητά τους να φέρουν εις πέραν το έργο τους. Το Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ να απορρίψετε το εναλλακτικό ψήφισμα που δεν εξυπηρετεί καθόλου τα συμφέροντα της δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κάσμαν. Να δώσω το λόγο στην κυρία Σουίτσα. Ευχαριστώ πολύ. Η εμπιστοσύνη των πολιτών είναι πολύ χαμηλή και γι' αυτό το λόγο η διαφάνεια χρειάζεται οπωσδήποτε. Αλλά από ό,τι ξέρω στις χώρες μέλη υπάρχουν νόμοι για το δικαίωμα στην πρόσβαση στην πληροφόρηση και αυτό το δικαίωμα προβλέπει ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να βλέπουν, να έχουν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, τα δημόσια έγγραφα. Αυτό ισχύει και για την Ένωση. Και ελπίζω ότι σύντομα θα είναι πράγματι δυνατόν οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε όλη την νομοθεσία της Ένωσης και θα, γνωρίζουν, θα μπορούν να γνωρίζουν πώς θα πανώνται τα χρήματα στην Ένωση. Μόνο έτσι θα υπάρξει πιο, πιο ενεργός ρόλος των πολιτών και μεγαλύτερη συμμετοχή τους. Και έτσι θα τους καλέσουμε πιο αποτελεσματικά να προσέλθουν και στα σκάλπας. Αυτό είναι ο σωστός τρόπος και γι' αυτό συμφωνώ ότι χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια. Ε, πρόεδρε, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και προφανώς στην Ευρώπη στην οποία ζούμε το κοινό δικαιολογημένα επιθυμεί περισσότερες πληροφορίες και θέλουν περισσότερη διαφάνεια και επιθυμούν καλύτερη πρόσβαση στα έγγραφα ε, και, ιδιαίτερα, και, να, ε, πραγματικά να τους τίθεν, δίδονται στη διάθεσή τους. Ε, και αυτό ισχύει τόσο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και για τα άλλα θεσμικά όργανα. Πολλοί συνάδελφοι ανέφεραν το ΕΛΚ. Εγώ δεν, εμένα δεν με αφορά άμεσα αυτό το θέμα, αλλά θέλω να υπάρξει μια διάκριση μεταξύ της πρόσβασης στα έγγραφα και της πρόσβασης στη διαδικασία. Προφανώς αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση και διαπραγμάτευση. Αλλά αν μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία στο σώμα αυτό εν σχέση με το τι είναι η διαφάνεια και κατά πόσο τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα ευχαρίστω στους πολίτες ανα πάσα στιγμή. Ευχαριστώ πολύ ο κύριο, η κυρία ο κύριος Πίτσουλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε εδώ πρέπει να διευκολύνουμε το έργο των ε, αρχών. Είναι πραγματικά προϋπόθεση για την καλύτερη επικοινωνία τους με τους πολίτες και για να είμαστε και εμείς αποτελεσματικότεροι. Να υπάρχει σωστή πληροφόρηση το δικαίωμα όλων των πολιτών που πρέπει να γίνεται σεβαστό. Ιδίως ό,τι αφορά την πρόσβαση σε έγγραφα, σε έγγραφα που ε, δεν είναι επιζήμια για τον ιδιωτικό τους βίο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά χωρίς να προκαλέσουμε ασαφής την, ισχύ, την ισχύ ασαφών κανόνων. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στην κοινωνία υπάρχουν ε, πολίτες με ψηλό ε, μορφωτικό επίπεδο, εκείνοι θα ενημερώνονται και θα λαμβάνουν τι σωστέ αποφάσει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα είναι διαφανέστερο και θα πρέπει να στηρίξουμε τη δημιουργία μια τέτοια κοινωνία. Πρόεδρο, ευχαριστούμε κυρία Τόμασιτ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ υποστηρίζω αυτή την έκθεση γιατί πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρξει συμβιβασμός για το θέμα της διαφάνειας. Η δουλειά των δημοσίων οργάνων, ο τρόπος που χρηματοδοτούνται, πρέπει να παρουσιάζονται ανοιχτά στο κοινό, στο οποίο είμαστε όλοι υπόλογοι. Αλλά είναι τραγική ηρωνία ότι το Κοινοβούλιο με έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας πάει να το κάνει, δύο εβδομάδες μόλις μετά που ψηφίσαμε την παράταση του ισχύω του άρθρου 147, καθυστερώντας έτσι την εφαρμογή του και για την Κροατία. Σε αυτή τη φάση οι Κροάτες έχουν πρόσβαση σε λιγότερο από το 50% των κειμένων στη γλώσσα τους. Γι' αυτό καλώ όλους τους διακεκριμένους συναδέλφους να σταματήσουν αυτή την άνηση μεταχείριση των Κροατών και να κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα και λοιπές πληροφορίες στη γλώσσα των. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Σόμερ. Κύριε Πρόεδρε, και το ΕΛΚ επιθυμεί διαφάνεια, πάντοτε είμαστε υπέρ της διαφάνεια, αλλά η διαφάνεια θα πρέπει να σταματάει εκεί που τίθεται σε κίνδυνο η προστασία των δεδομένων. Στην ε, έκθεση ε, αναφέρεται αυτό το οποίο ζήτησε και ο κύριος ε, Κάσμαν εδώ και πολλά χρόνια. Και χαίρομαι κύριε Κάσμαν που θα εγκαταλείψετε το κοινοβούλιο και ίσως έτσι προχωρήσουμε περισσότερο εμείς οι υπόλοιποι. Ε, συγχαίρεται την πρόσβαση στα έγγραφα με την πρόσβαση στη διαδικασία. Και ναι, η νομοθετική διαδικασία είναι σύνθετη, είναι πολύπλοκη και πράγματι υπάρχει μια φάση την οποία δεν μπορεί να δημοσιοποιεί κανεί ανα πάσα στιγμή. Για παράδειγμα στο επίπεδο των ε, τριλόγων. Εάν κυρία Συγήτρια είχατε συμμετάσχει ε, σε κάποιο τρίλογο θα βλέπατε ότι δεν είναι δυνατή η πρόσβαση του κοινού στα δημόσια έγγραφα σε αυτή ακριβώς τη φάση. Ε, δεν δυνατόν να αποκαλύπτεται εσωτερικά ε, διοικητικά στοιχεία ή διάφορα δεδομένα περί ανταγωνισμού. Έχετε, γύρετε την αξίωση της απολυτότητας. Ε, δεν επιθυμείτε να συνομιλήσετε με το ΕΛΚ. Αντίθετα, επηρεαστήκατε από τον συνάδελφο κύριο Κάσμαν. Ε, γι' αυτό ε, το ΕΛΚ συνέταξε ένα δικό του ψήφισμα που κατά την άποψή μας ε, συνοψίζει καλύτερα την κατάσταση. Κυρία, κυρία Σόμερ μου, θα έχετε μία ερώτηση από την κυρία Ιντεφέλντ. Δέχομαι. Ορίστε. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι δεν είμαι ικανοποιημένο που φεύγει ο κύριος Κάσμαν μετά από όλα όσα έκανε εδώ μέσα μετά από 15 χρόνια δεύτερον έχω συνοηθεί με το ΕΛΚ και υποστήριξα πολλές από τις εξαιρετικές του τροπολογίες όπως της κυρίας Κοράτσα Μπίλντα αλλά ερωτώ δεν πιστεύετε ότι οι ίδιοι οι πολίτες είναι οι καλύτεροι κριτές του τι πληροφόρηση πρέπει να και θέλουν να έχουν και τι να μην έχουν. Γιατί αρνείστε αυτού του είδους το άνοιγμα δεν σημαίνει ότι όλα θα είναι προσβάσιμα αλλά προς στιγμήν η μυστικότητα φαίνεται να είναι ο κανόνας. Έχω και άλλη εμπειρία με τριμερείς διαλόγους και με δικαστήρια ως προς τη διαφάνεια. Εσείς έχετε τέτοια εμπειρία κυρία Σόμερ. Παρακαλώ απαντήσατε. Κυρία συνάδελφε, εδώ και 15 χρόνια είμαι μέλος αυτού του κοινοβουλίου και έχω διαπραγματευτεί σε πολύ δύσκολους ε, τριλόγους για πολύ επίμαχα θέματα και με έντονη συμμετοχή των ομάδων λόμπι. Γι' αυτό γνωρίζω πολύ καλά περί την ομιλώ. Ε, ναι, γιατί δεχτήκατε κάποιες τροπολογίες ε, του ΕΛΚ από την κυρία Κοράτσα Μπίλτ για παράδειγμα επειδή συμφωνούν με τη δική σας άποψη, αλλά δεν ασχοληθήκατε καθόλου με άλλες τροπολογίες του ΕΛΚ γι' αυτό ισχύει το ότι γύρεται μια αξίωση απολυτότητας αλλά ε, δεν είσαστε οι μόνοι που έχετε το προνόμιο της σοφίας ε, βεβαίως μπορεί κανείς ε, να αποκαλύψει πολλά πράγματα, αλλά όχι τα πάντα και εν πάση περιπτώσει όχι εσείς επιθυμείτε να αποκαλύπτονται. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον κύριο Μπόρκ ε, για να καταλήξει. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι βουλευτές, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Ινθβέλ, που μίλησε για τη ζωτική σημασία της αρχής της διαφάνειας και της δημοκρατικής συμμετοχής ως προς την λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Βεβαίως, είναι κοινή ευθύνη του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής να διασφαλίσουν το απαραίτητο επίπεδο διαφάνειας στη λειτουργία των ε, ε, θεσμικών οργάνων. Και αυτή η ευθύνη έχει να κάνει και ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στο ε, τομέα της διαφάνειας, την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα που καλύπτεται από το σχετικό κανονισμό με ακριβώς αυτό το τίτλο. Ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός εγγράφων στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση είναι κάτι που έχουν ζητήσει και οι Ευρωπαίοι πολίτες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με 6.000 αιτήσει πρόσβαση ετησίω. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτε διαρκώ ε, συνειδητοποιούν τα δικαιώματά του στον τομέα αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ικανοποιήσει πάρα πολλά από τα αιτήματα που έχει λάβει για την πρόσβαση στα έγγραφα. Περισσότεροι από περισσότερα από 4 στα 5 αιτήματα ε, ικανοποιούνται στο πρώτο στάδιο. Και η είναι περίπου 200 οι αιτήσει μόνο που απορρίπτονται ετησίω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να ε, υλοποιήσει και έχει όντω ανταποκριθεί σε αυτή την υποχρέωση να ικανοποιεί διαρκώ, να, σε, να εφαρμόζει μάλλον διαρκώ συστηματικά και αποτελεσματικά την αρχή αυτό. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο άλλωστε έχει ελέγξει την συμμόρφωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υποχρέωσή τη έχει δώσει μεγάλο, μεγάλο έμφαση στους τριμερούς διαλόγους η συγκύτρια. Για τους τριμερούς διαλόγους όντως και ε, ο συνομοθέτης έχει ευθύνη για να ε, ορίσει το κατάλληλο επίπεδο διαφάνεια στον τομέα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φροντίζει πάντως τα κείμενα που δημοσιεύονται να είναι εύληπτα, ισόρροπα και ενημερωτικά. Ε, θα πρέπει όμως να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ του σωστού επίπεδου διαφάνειας και της ε, σκόπιμης νομοθετικής δράσης. Θα πρέπει να συντάσσουμε έγγραφα τέτοια που να είναι περισσότερο συγκρίσιμα και να είναι ακριβώς ε, δυνατή η πρόσβαση σε αυτά. Ως προς τις δικές σας ε, μέρημνες για τον κανονισμό αυτό παραμένουμε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε και τα δύο κεφάλαια, τα δύο βασικά κεφάλαια και τους δύο βασικούς πυλώνες της ε, τρέχουσας πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστούμε κύριε Μπόρτς. Η συζήτηση κλείνει, η ψηφοφορία αύριο στις 12. Τώρα, επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, έκθεση έκθεση του κυρίου Βαλέσα, δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2013. Να δώσω τον λόγο στον εισηγητή.